We, our group was uh, people. Ex- no, that's right. Um, our group was um, people. People, let's do it. All right, I'll give it a try. Ε, το, η ομάδα μας ε, ασχολήθηκε με τα, με τα άτομα τα οποία ήταν, ε, είναι γενικά ε, εκτός της κοινωνίας λόγω κάποιων ε, προβλημάτων ε, που έχουν, ε, είτε λόγω προβλημάτων λεφτών που είναι σε αυτήν την κατηγορία poverty όπως το, όπως το συζητήσαμε είτε με προβλήματα κινητικότητας είτε με διαφορετικό γένος. People are looking at me with weird looks. Me, you are speaking too loud uh, compared to what you are here. Okay, speaking okay, I'm speaking Greek. I, speak in English. Uh, so um, our group was people excluded